Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε σημείο 14. Πιλωτικά σχέδια για την νόμιμη μετανάστευση, τρέχουσα κατάσταση. Δεν έχω μαζί μου τα γυαλιά μου, αν και δεν νομίζω ότι θα εντυπωσιάσει κανένα αυτό. Εμένα όμως μου δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο λοιπόν, Μετανάστευση 2015 δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσα να κάνω μια πολύ μακρά παρουσίαση, αλλά έχουμε την κυρία Μίχο, τη Γενική Διευθύντρια, η οποία θα έπρεπε να έχει έρθει, όμως δεν μπορεί την εκπροσωπεί ο συνάδελφός της από τη Γενική Διεύθυνση. Έχει καθυστερήσει μια στο Συμβούλιο, κυρία Μίχο. Θα μας κάνετε λοιπόν μια παρουσίαση για τα πιλωτικά προγράμματα, για την σχέδια για την νόμιμη μετανάστευση και μετά θα γίνει συζήτηση. Παρακαλώ, Ματσίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ξέρετε, η Επιτροπή εδώ και αρκετό καιρό επιδιώκει την προβολή της ε, διαχείρισης της μετανάστευσης ε, την αντικαταστήση και την αντικατάστασή της από την νόμιμη. Να μην μιλούμε μόνο για διαχείριση δηλαδή μετανάστευση αλλά από νόμιμη μετανάστευση και θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημαντικά εργαλεία τα οποία υπογραμμίζουν την προσέγγιση καταρχάς την ε, ανακοίνωση για την νόμιμη μετανάστευση του Σεπτεμβρίου 2018 και δεύτερον την τελευταία έκθεση προόδου για το θεματολόγιο για τη μετανάστευση της 9 Δεκεμβρίου του 2018. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την ιδέα για πιλωτικά σχέδια για την μετανάστευση το Σεπτέμβριο του 2017. Από κοινού με τα κράτη-μέλη που θέλησαν να συνεργαστούν, 14 τον αριθμό, σχεδιάσαμε αυτά τα κοινά πιλωτικά σχέδια περιγράψαμε το, την, κοινή, την ιδέα, την οποία άλλωστε το Μάρτιο του 2018 παρουσιάσαμε στην Επιτροπή σας. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είχαμε εξ αρχής ε, εντατικές ανταλλαγές με διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς οικονομικούς φορείς ε, Παγκόσμια Τράπεζα, BERD, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, και ICNPD και στόχος ήταν να εξασφαλίσουμε κοινέ αξίες και συνεργατικές σχέσεις. Οι διεθνείς αυτοί φορείς λοιπόν, όπως ξέρετε, ίσως είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν και την εφαρμογή των σχεδίων αυτών. Έχει εκφραστεί γενικά υποστήριξη λοιπόν στην ιδέα αυτή των πιλωτικών σχεδίων και θα θέλω να τονίσω ότι με τα πιλωτικά σχέδια για την νόμιμη μετανάστευση καταθέτουμε ως Επιτροπή και ένα συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά και υποστήριξη χρηματοδότησης που διαθέτουμε ήδη στα κράτη-μέλη που είναι διτεθειμένα να ξεκινήσουν την εφαρμογή των σχεδίων. Πολύ σύντομα θα ήθελα να εξηγήσω ποια είναι η ιδέα αυτή των πιλωτικών σχεδίων με μια πολυσχεδή στρατηγική. Θέλουμε λοιπόν ε, αυτή η στρατηγική που θα είναι υποφελής για όλους ε, να σχεδιαστεί για τα κράτη-μέλη. Κράτη-μέλη τα οποία έχουν και δημογραφικά προβλήματα και ανάγκες για ενσωμάτωση στις ε, χώρες, αγορές εργασίας των μεταναστών, τη δυνατότητα για πρόσληψη έστω και προσωρινά μεταναστών από αφρικανικές χώρες. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια εποφελή για τα κράτη αυτά κατάσταση και να χορηγήσουμε, θέλω να το τονίσω αυτό, τη μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν μόνο τους να ορίσουν τα ορόσημα και τα κριτήρια για αυτά τα σχέδια. Θέλουμε να είναι επωφελής όμως και για τους μετανάστες η κατάσταση αυτή, καθώς αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξασφαλίσουν την κατάρτιση, να εργαστούν σε επιχειρήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα όταν θελήσουν να επαναπατριστούν, να έχουν και το κίνητρο υποφελούμενος εκ τούτου από την υποστήριξη ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα τους επιτρέπουν παραδείγματι να ε, ιδρύσουν μια επιχείρηση στη χώρα τους. Και κάτι ακόμη, εποφελές θα είναι το σχέδιο αυτό και για τις χώρες προελεύσεως. Καταρχάς, γιατί με την προσωρινή αυτή μετανάστευση αποφεύγουμε τον brain drain ει βάρος των κρατών προελεύσεω, κάτι το οποίο συχνά επικρίνεται. Δεύτερον, οι επανερχόμενοι στις αιστείε τους αυτοί οι μετανάστες θα δημιουργούν θέσει εργασία, ιδρύοντας νέες επιχειρήσεις και οι χώρες προελεύσεως επίσης θα μπορούν να επωφεληθούν από τις δεξιότητες και γνώσεις που θα έχουν εντωμεταξύ αποκτήσει οι ε, πολίτες τους. Αυτή είναι η βασική ιδέα λοιπόν. Προς το τέλος ε, του 2018 είδαμε συγκεκριμένα σχέδια από ορισμένα κράτη-μέλη που τώρα έχουν ετοιμαστεί λίγο πολύ και μπορούμε να πούμε ότι τα πιλωτικά σχέδια εξελίσσονται προς την ορθή κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, το Βέλγιο και η Λιθουανία ήταν τα πρώτα που ε, έκαναν ε, προτάσεις για το σχέδιο κινητικότητας και εταιρικής σχέσης ε, σε σχέση με το, με το Μαρόκο και την Ιγυρία Αντιστοίχω, με προαγωγή της νόμης μετανάστευσης σε πιλωτικό στάδιο ε, βραχυπρόθεσμα και μέσοπρόθεσμα. Ε, πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με την στόχευση να μην εγκαταλείψουν τη χώρα προελεύσεως οι μετανάστες ή να τους ενθαρρύνουν να επανέλθουν στις πατρίδες τους προκειμένου να δημιουργήσουν, όπως είπα, τη δική τους επιχείρηση. Και άλλα σχέδια αναπτύσσονται από άλλα κράτη-μέλη που στόχο έχουν κυρίως χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ταυτόχρονα όμως προάγουμε και την ιδέα της ε, ε, δραστηριοποίησης και στο χώρο της, νο... της νοτίως της Σαχάρας Αφρικής. Εδώ έχουμε κυρίως τη Γερμανία αλλά και το Βέλγιο, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Πρωτοβουλίες που συνεχίζονται και σχεδιάζονται περαιτέρω και έτσι προχωρούμε περισσότερο στις, ε, στην πτυχή της συνεργατικής δράσης. Όταν στην ίδια τρίτη χώρα ενδιαφέρον έχουν δείξει περισσότερες χώρες πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργατική σχέση, τουλάχιστον η αμοιβαία αντίληψη ότι υπάρχουν οι δραστηριότητε των ΜΕΝ και των ΔΕ και γι' αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρώτο τρίμηνο του 2019 οργανώνει workshop, εργαστήρια ενημέρωση σε σχέση με τι χώρε τη Βόρειας Αφρική, για να έχουμε καλύτερο συντονισμό και συνεργατική σχέση που μπορεί οπωσδήποτε να αναγνωριστεί ω πολύ καλό στόχο για τέτοιου είδου σχέδια στο χώρο τη πολιτική και για την ανάπτυξη. Πρόεδρε, σταματώ εδώ. Πολύ ευχαριστώ απαντήσω στις ερωτήσεις των βουλευτών. Ευχαριστώ πολύ. Η Τζούντιθ Σαρτζεντίνη. Α, γρήγορα τα είπατε. Ακούγοντας σας, δεν ξέρω κατά πόσο μιλάμε για τους οικονομικούς μετανάστες ή θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για τις ε, έρευνες σε σχέση με τα σχέδια ιδιωτικού ευρωπαϊκών ε, χορηγιών και υποστηρίξεων. Τώρα, σε σχέση με τα προγράμματα ε, μετανάστευσης που σκιαγραφίσατε, βλέπω ότι μιλάμε και για ε, επαναπατρισμούς, γιατί αν μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες ως εργατικό δυναμικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εργοδότες θέλουν να έχουν εργαζομένους προς εκπαίδευση, αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι όταν αποχωρεί αυτός ο εργαζόμενος. Δεν έχει νόημα λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας στην κατάρτιση και εκπαίδευση και μετά επιστροφή θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για άλλα προγράμματα τα οποία δεν είναι κυκλικά. Γιατί έτσι δεν θα, δεν θα έχει νόημα να μιλάμε για μετακινήσεις όπου κανείς επαναπατρίζεται. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και να επανέλθει. Επίσης, ποιο είναι το επίπεδο κατάρτισης που ζητάτε, για τι εργασία μιλάμε. Μιλάμε και για εργασίες ε, για ε, χαμηλές ηλικίες, γιατί πολλοί ε, παράνομοι μετανάστες καταλήγουν σε εργασία που απασχολεί ε, άτομα μικρής ηλικίας και βέβαια που κακοπληρώνονται. Ε, ο κύριος Διούρεκα, ε, ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο μου ερώτημα έχει ως εξής. Ε, ποια είναι τα αριθμητικά στοιχεία για τους νεοεισερχόμενους που αναμένετε στα προγράμματά σας. Και το δεύτερο, τα προγράμματα αυτά είναι άκρος ενδιαφέροντα, αλλά μιλάμε και για εκείνους οι οποίοι θα επανέλθουν, θα επιστρέψουν στη χώρα τους για να δημιουργήσουν εκεί μια επιχείρηση και για να δημιουργήσουν ένα νέο δυναμικό και μια δυναμική για αυτές τις χώρες. Νομίζω ότι η Επιτροπή έχει κάνει τέτοιους υπολογισμούς. Κάποιος άλλος. κυρία Σαρτζεντίνη ε, μίλησε για, την, για το γεγονός ότι η παρουσίαση ήταν πολύ περιορισμένη, είναι πολύ περιορισμένη. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες ε, αυτών των σχεδίων επί του παρόντος και ως προς την γενικότερη πολιτική και τις προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου της έχουμε και την οδηγία για την μπλε κάρτα που έχει υποβάλει η Κομισιόν στο Συμβούλιο. Εγώ θα ήθελα να υποβάλω ε, το εξή ερώτημα. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί ε, γιατί το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς την νόμιμη μετανάστευση και τους ε, διαδρόμους που δημιουργούνται για αυτή την νόμιμη μετανάστευση. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής. Εσείς ε, θεωρείτε ότι πρέπει να προβάλλετε προγράμματα ιεραρχικά ε, βαθμιαία δηλαδή με βάση και τις ε, δημογραφικές ανάγκες και ανάλογα με το μέγεθος του προγράμματος ή είσαστε πιο φιλόδοξοι γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ κακή περίοδο ως προς την ε, νόμιμη μετανάστευση αν μιλήσω ως εισηγητής για την μπλε κάρτα και γιατί ακριβώς γίνεται λόγος και για πάγωμα της ε, νόμιμης μετανάστευσης με αυτά τα μέτρα που λαμβάνετε. Πώς βλέπετε τα πράγματα. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα χάσμα, θα το αφήσετε για αργότερα ή θα μιλήσετε για αυτούς τους νόμιμους διαδρόμους που είναι απολύτως απαραίτητοι. Ευχαριστώ. Κύριε Μωράης, θα αρχίσουμε τη δική σας ερώτηση γιατί αφορά το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Η Επιτροπή ε, λυπάται ιδιαίτερα γιατί δεν θα υπάρξει πολιτική συμφωνία για τη μπλε κάρτα κατά τη θητεία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τη δική μας πλευρά καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ε, για να προωθήσουμε το θέμα. Θα μπορούσα να πω ότι αν λάβουμε υπόψη ότι τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται την αγορά εργασίας και τα κοινωνικά συστήματα, υπάρχει ε, μετανάστευση η οποία είναι κυρίως παράνομη και όχι τόσο νόμιμη. Μετά το 2015 μπορούμε να πούμε ότι και άλλα ζητήματα ανέκυψαν σε σχέση με την διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης Άρα το θέμα αυτό δεν ήταν προτεραιότητα για το Συμβούλιο. Θα αναφερθώ στην ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νόμιμη μετανάστευση. Νομίζω ότι υπάρχει πολιτική συμφωνία παντού, διαθεσμικά δηλαδή, ότι θα πρέπει να περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το μέγιστο δυνατό. Αυτή είναι η πολιτική πρόθεση όλων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε εκεί. Εάν περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση θα πρέπει να την αντικαταστήσουμε με την νόμιμη τακτική μετανάστευση και εδώ Μπαίνουν και οι ε, μπλε κάρτες, εδώ εντάσσονται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει έλεγχο καταλληλότητας για την νόμιμη μετανάστευση. Ε, πρόκειται για ένα fitness check το οποίο θα ε, οδηγήσει σε συμπεράσματα που θα υποβληθούν έτσι ώστε να γίνει δημόσια διαβούλευση και συζήτηση για την νόμιμη μετανάστευση έτσι ώστε κατά την επόμενη θητεία να φτάσουμε σε μια συνεκτική προσέγγιση για την νόμιμη μετανάστευση γιατί δεν μπορούμε απλώς να πούμε ότι πρέπει να σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση. Θα πρέπει να δούμε το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης προς την αγορά εργασίας και το θέμα, τα θέματα βέβαια επαναπατρισμού εκεί που υπάρχουν. Το ερώτημα της κυρίας Αργεντίνη τώρα. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι αν λάβουμε υπόψη το ότι το θέμα αυτό είναι ευαίσθητο, βλέπουμε αυτά τα ε, πιλωτικά σχέδια σαν ένα πείραμα Γι' αυτό ε, τα κράτη-μέλη έχουν ευελιξία ως προς το σχεδιασμό για να δουν τις ανάγκες και δεν θέλουμε να πιέσουμε με αριθμητικά στοιχεία. Θέλουμε να μπει σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο και 12 κράτη-μέλη μέχρι τώρα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτά τα πιλωτικά σχέδια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν μιλάμε για τη μετανάστευση προς την αγορά εργασίας, αλλά μπορούν να καλυφθούν και οι φοιτητέ. Αυτό αφορά το ισπανικό πιλωτικό σχέδιο, το οποίο τώρα βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας και ως προς τις ιδιωτικές χορηγίες, εδώ μιλήσατε για ένα ξεχωριστό ζήτημα οι ιδιωτικές αυτές χορηγίες βρίσκονται στο στάδιο μελέτης και υπάρχει ένα πιλωτικό σχέδιο της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χορήγησης Ασύλου. Θα πρέπει να γίνει αυτή, αυτός ο διαχωρισμός των ιδιωτικών χορηγιών και επιδοτήσεων και το θέμα της μετανάστευσης. Επίσης, δεν ορίζουμε το επίπεδο εκπαίδευσης σε αυτά τα πιλωτικά. Μιλάμε για ανθρώπους που θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή κατάρτιση, αλλά χρειάζεται και νοσηλευτικό προσωπικό και ούτω καθεξής. Ως προς τα αριθμητικά στοιχεία για μας τα στοιχεία αυτά δεν είναι τόσο σημαντικά ως, προ, ως ε, προς το γεγονός ότι τα πιλωτικά προγράμματα θα πρέπει να καταστούν ε, λειτουργικά. Για τη Λιθουανία έχουμε 59 Νιγηριανούς, για το Βέλγιο 60 Μαροκινοί θα συμμετάσχουν και για τα άλλα πιλωτικά σχέδια δεν έχουμε όλα τα αριθμητικά στοιχεία. Από πλευράς όμως ε, επιτροπής ε, σημασία έχει η δοκιμή και όχι ο αριθμός συμμετεχόντων για να δούμε κατά πόσο θα υπάρχει ένα λειτουργικό πλαίσιο έτσι ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη. Γι' αυτό δεν έχουμε και υπολογισμούς για το οι μετανάστες θα επαναπατριστούν. Υπάρχουν πιλωτικά σχέδια. Συμφωνώ με την κυρία Σαρτζεντίνη ότι φυσικά οι εργοδότες θέλουν να κρατήσουν καλό προσωπικό εκεί που υπάρχει. Αλλά αυτό ε, έχει σχέση και με τη χρηματοδότηση και εκεί υπάρχουν κίνητρα επιστροφής ή όχι. Υπάρχει μια κρίσιμη μάζα συμμετεχόντων όταν οι εργοδότες δεχτούν να υπάρξει τουλάχιστον μία προσωρινή βάση εφαρμογής. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Με την δημοσίευση του fitness check της ε, νόμιμης μετανάστευσης θα έχουμε το επόμενο βήμα που θα μας δώσει μια επισκόπηση των εξέλιξεων. Ευχαριστούμε πολύ που μας ενημερώσατε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τους ε, συναδέλφους που έθεσαν ερωτήσεις. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Αν είμαστε όλοι εδώ και έτοιμοι.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 να ζητήσουμε τον κύριο Νέτσι να έρθει πιο νωρίς για το τελευταίο ζήτημα, έτσι ώστε να τελειώσουμε συνολικά νωρίτερα. Κανένα δεν νοιάζεται που εγώ προσπαθώ να συντομεύσω τη συνεδρία, σε ό,τι φαίνεται. Τέλο πάντων, εγώ θα επιμείνω. Okay. Hello. So, colleagues, um, Άμεσα συνδεόμενο με το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης είναι η ένταξη. Είναι το ζήτημα της ένταξης, το, στο οποίο εμείς επιμένουμε. Είχαμε και μια πολύ καλή εμπειρία εκθέσεων και briefings από το ελεγκτικό συνέδριο. Η διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών πρόσφατα ανέλησε μια έκθεση για το αντίκτυπο των εκθέσεων του Συμβουλευτικού Συνεδρίου στο έργο της Επιτροπής μας αλλά και στο έργο άλλων επιτροπών. Και χαιρόμαστε που ο αντίκτυπος αυτός είναι σημαντικός. Ε, σήμερα έχουμε μια έκθεση για την ένταξη των μεταναστών είναι ένα ενημερωτικό έγγραφο που εστιάζεται πιο πολύ στη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα άλλο, μια κοινή δημοσίευση με τον ΟΣΑ, μεταξύ ΟΣΑ και Γενική Διεθνή Home, ε, για, συνολικά για τι χώρε του ΟΣΑ και του G20, ε, για του ε, δείκτες περί 74 συνολικά δείκτες για την ένταξη των μεταναστών. με τις τρεις πυρώνες, η αγορά εργασίας, ε, συνθήκες διαβίωσης και κοινωνική ένταξη. Η ένταξη των μεταναστών είναι προφανώς ε, κύρια ευθύνη των κρατών μελών, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει και αυτή σημαντικό ρόλο με κίνητρα και στήριξη. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αλλά και χρηματοδότηση για πολιτικές ένταξης και αποφύγης των διακρίσεων. Οπότε πρώτα θα μας μιλήσει η κυρία Ιβάνοβα, που είναι υπεύθυνη για το ενημερωτικό έγγραφο αυτό του ε, Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για 10 λεπτά. Μετά θα ακούσει ερωτήσεις. Όχι, όλες μαζί ερωτήσεις. Οκ. Okay. Κάποιοι θα φύγουν νωρί. Ε, δεν χρειάζεται να φύγει τελικά νωρί, γιατί αρχίσαμε νωρί. Πάση περιπτώσει. Τι εννοούσα. Εννοούσα ότι όλοι να μείνετε εδώ και να μην φύγει κανένα. Αυτό εννοούσα. Και μετά θα πάρει το λόγο και ο Στέφανος Καρπίστα του ΟΣΑ. Σας προειδοποιώ για αργότερα κύριε Σκαρπίστα. Και θα δώσουμε το λόγο επίσης και σε ένα εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Home. Για 10 λεπτά συνολικά. Λοιπόν, ο λόγος στην κυρία Ιβάνοβα καταρχήν. Ενημερωτικό έγγραφο του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Πάντα χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλο ότι η παρουσία μου είναι η πρώτη μου παρουσία σε αυτή την Επιτροπή. Συνήθως συζητώ θέματα συνοχής. Όπως είπατε όμως αυτή τη φορά μιλάμε για την ένταξη των μεταναστών. Είμαι υπεύθυνη για αυτό το ζήτημα, οπότε με χαρά μου θα σας παρουσιάσω αυτό το θέμα σήμερα να συγχαρώ και τους συναδέλφους του ΟΣΑ και της Επιτροπής ε, για τη δική τους ε, λεπτομερή μελέτη περί των δικτών ένταξης των μεταναστών. Μία από τις προκλήσεις, οποίες έτσι κι αλλιώς εμείς ε, εντοπίσαμε στο δικό μας ενημερωτικό έγγραφο, είναι η ανάγκη να έχουμε μια αποτελεσματική παρακολούθηση του αποτελέσματος των, πολιτικών, των ενταξιακών μας πολιτικών, προκειμένου αν χρειάζεται να προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας. Να σας υπενθυμίσω ότι το έγγραφό μας δημοσιεύτηκε τον περασμένο Μάιο, το οποίο σημαίνει ότι η ανάλυση μας είναι λίγο παλαιότερη από τα δεδομένα τα οποία θα σας παρουσιάσουν αργότερα οι επόμενοι ομιλητές. Η πρόσφατη αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζητούν προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έφερε την μεταναστευτική πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των συζητήσεων ε, τα έτη 2014-2017, τέσσερα χρόνια, 3,7 εκατομμύρια περίπου άτομα ζήτησαν άσυλο για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τέσσερα αυτά χρόνια, τρει φορές περισσότεροι από ό,τι την προηγούμενη τετραετία. Μπορείτε να δείτε εδώ το, τον τύπο των ατόμων τα οποία ε, στα οποία αναφερόμαστε ε, δεν συμπεριλαμβάνουμε τα άτομα τα οποία παραμένουν παρανόμως στις χώρες, στα κράτη-μέλη. Γιατί εκεί υπάρχει, υπάρχουν ειδικέ εκθέσεις οι οποίες αφιερώνονται σε αυτούς και οι οποίες θα δημοσιευθούν σε λίγο καιρό. Εδώ βλέπουμε πού ακριβώς λαμβάνει η χώρα η ένταξη. Είναι ένα από τα βήματα της διαδικασίας μετανάστευσης, ε, της ε, διαδρομής μετανάστευσης. Ε, ξεκινάμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός των συνόρων μας, μετά έχουμε τον έλεγχο των συνόρων και την υποδοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά η ένταξη, η οποία μπορεί να δώσει πολλά μακροπρόθεσμα ωφέλη στις χώρες στις οποίες γίνεται αυτή η ένταξη, όπως έχει αποδειχθεί από τις μελέτες. Η ένταξη των μεταναστών στις ε, κοινωνίες αποτελεί βασική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει κίνητρα και να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη σε αυτό τον τομέα. Πλευρά χρηματοδότηση έχουμε διάφορα εργαλεία, διάφορους διάβλους μέσω των οποίων ε, κονδύλια φτάνουν στα κράτη-μέλη. Παρόλο ότι δεν είναι εύκολο εύκολο να εντοπιστεί ποιο είναι το ακριβές ποσό το οποίο αφιερώνεται στην ε, ένταξη, στις δράσεις των διαφόρων ταμείων ή των διαφόρων εργαλείων που διαθέτουμε. Τώρα, τι είναι η ένταξη, δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω, αλλά αυτή είναι μια, ε, ε, μια περιγραφή των βασικών δράσεων και των βασικών αρχών της ένταξης. Ε, περιλαμβάνεται, περιλαμβάνεται στο νούμερο 3, όπως βλέπετε, η απασχόληση, έχουμε τη στέγαση, έχουμε την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει επίσημος ορισμός ε, της ένταξης. Ε, στο, το 2004 αυτές οι 11 βασικές αρχές, οι οποίες βλέπετε εδώ, θεωρούνται ε, σημαντικές ε, και περιέγραφαν το φαινόμενο της και το περιγράφουν ακόμα και τώρα. Όπω και τα περισσότερα προϊόντα του ελεγκτικού συνεδρίου, αυτό το ενημερωτικό έγγραφο δεν είναι μια επίσημη έκθεση, παρόλο ότι ακολουθούμε αυστηρά κριτήρια και στα ενημερωτικά μα έγγραφα. Συνεπώ ε, τα, ο, ο στόχος του είναι να πυροδοτήσει μια πολιτική συζήτηση για αυτό το θέμα. Οπότε, περιγράφει και συνοψίζει τις δράσεις των κοινοτικών οργάνων σε θέματα ένταξης με ιδιαίτερη εστίαση στις αντιδράσεις που προέκυψαν στην αντίδραση των κρατών μελών στο, στην αύξηση των μεταναστευτικών οργών. Πέντε ήταν, ε, εφτά ήταν οι προκλήσεις οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν οι πολιτικές ένταξης, ε, τις οποίες εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη και που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σας είπα. Πάντω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει ρόλο συμβουλευτικό έτσι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε θέματα ένταξη των μεταναστών. Ποιε είναι αυτέ οι προκλήσει λοιπόν. Πρώτη πρόκληση. Η μείωση των καθυστερήσεων στην έναρξη της διαδικασίας ένταξης. Η εφαρμογή του μεταναστευτικού δικαίου είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών καταρχήν βέβαια, γιατί μεταγράφουν την ε, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία και τα κράτη-μέλη έχουν την ευχέρεια, τη διακριτική ευχαίρεια να το κάνουν αυτό, αυτή τη να την κάνουν με διαφορετικούς τρόπους, γι' αυτό λόγο ισχύουν και ελάχιστα διαφορετικοί κανόνες. Ε, και αυτές οι διαφορές μπορούν να οθήσουν τους μετανάστες να μετακινηθούν από τη μια χώρα σε άλλη. Το 2016 το 30% των ετούντων άσυλο είχαν ήδη καταθέσει αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό βέβαια δημιουργεί καθυστερήσει στην έναρξη της διαδικασίας ένταξης ε, και ε, προφανώς δυσκολεύει την ένταξη. Ένας άλλος παράγοντας είναι η περίοδος αναμονής για την επεξεργασία των αιτήσεων. Οι διαδικασίε είναι πολλές φορές αργές και καθυστερούν. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση. Δεύτερη πρόκληση, το να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα ίδια δικαιώματα και την έλλειψη των διακρίσεων για όλους σημαντικός στόχος αυτό για να βοηθήσουμε τους μετανάστες να ενταχθούν. Στην ε, έρευνά μας τέσσερα κράτη-μέλη δήλωσαν ότι ε, η νοοτροπία του ντόπιου πληθυσμού έναντι των μεταναστών έχει, αρνητική, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ένταξή τους. Και πρέπει να γίνονται προσπάθειες για να αποφεύγονται οι διακρίσεις. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2017, περισσότερο από το 50% των Ευρωπαίων έχουν αρνητική αντίληψη για τους μετανάστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν ΔΕ, χρειάζεται να βελτιωθεί αυτή η νοοτροπία και να εξασφαλιστεί καλύτερη πρακτική εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ε, υπεθυμίσει τη σημασία του ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ένταξη των μεταναστών. Τρίτη πρόκληση που έχει σχέση με τη χρηματοδότηση και την αξιολόγηση των αναγκών, την εκτίμηση των αναγκών. Ε, κατόπιν της ε, αύξησης της μετανάστευσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια πρόσθετους πόρους για τη μετανάστευση. Ε, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς τους πόρους ε, αφιερώθηκε στην ε, ένταξη. Το, τα ποσά είναι ψηλά, αλλά το ΆΜΙΦ, ε, που είναι το Ταμείο για τη Μετανάστευση, δεν ε, καθιστά τελείω απόλυτα σαφέ ποιο είναι το ποσό το οποίο τελικά δαπανήθηκε για την ένταξη από τα κράτη-μέλη. Ούτε και τον αριθμό των μεταναστών που ήταν δικαιούχοι. Γι' αυτό το λόγο δεν κάναμε και πλήρη έλεγχο απόδοσης. Και είναι μόνο ένα ενημερωτικό έγγραφο αυτό που σας παρουσιάζουμε. Ε, γιατί τότε που έγιναν αυτές οι, που κάναμε αυτή την εξέταση ε, δεν είχαμε δεδομένα. Τα κράτη-μέλη όμω είπαν ότι στην ενδιάμεση, κατά τη διάρκεια τη ενδιάμεση αξιολόγηση του Ταμείου είπαν ότι χρειάζονται περισσότερα, μεγαλύτερα ποσά. Και σίγουρα είναι απαραίτητο να γίνει μια συνολική αξιολόγηση των αναγκών και τη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να ε, τεθούν στη διάθεση των κρατών μελών τα κατάλληλα ποσά, την, το κατάλληλο χρονικό, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να συμπληρώσει την, ε, ε, την ε, πολιτική ε, των κρατών μελών, γιατί αλλιώς μπορεί τα πράγματα, η πολυδράση μας να μην είναι αποτελεσματική. Τέταρτο, τέταρτη πρόκληση, η προσήλωση των κρατών μελών στην εφαρμογή του προγράμματος δάσης κομισιών. Η Κομισιόν λαμβάνει έτσι ένα συντονιστικό ρόλο σε θέματα ένταξης ε, στα μέτρα πρώτης ε, αποχώρησης, στην άφηξη, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας. Και αυτό το πρόγραμμα δράσης ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εστιάσουν στα πρόσθετα εθνικά μέτρα που μπορούν να λάβουν. Όμως αυτά τα μέτρα δεν θα τα παρακολουθεί η Κομισιόν, οπότε δεν θα μπορέσει να δώσει περισσότερη στήριξη στα κράτη-μέλη. Πέμπτη πρόκληση είναι η στήριξη όλων των μεταναστών σε όλες τις διαφορετικές σχετικές πολιτικές. Δηλαδή, κάποια κράτη-μέλη έχουν εθνικές πολιτικές ε, ε, ένταξης, άλλα αναπτύσσουν δράση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, άλλες χώρες ε, συμπεριλαμβάνουν τους μετανάστες σε διάφορες πολιτικές, όμως πολλές φορές κάποια κράτη-μέλη δεν λαμβάνουν ειδικέ δράσεις για νέους ή για απάτριδες ή για κάποιους τομείς της ένταξης, όπως για παράδειγμα η στέγαση ή η απασχόληση. Ε, και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια επίσης εντόπισαν συγκεκριμένες αδυναμίες σε ό,τι φορά τις πολιτικές των κρατών μελών για την ένταξη. Για παράδειγμα, ορισμένα μέτρα δεν ε, ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγκες των μεταναστών ή ε, για παράδειγμα η προστασία περιορίζεται στην πρωτεύουσα μόνο και όχι σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια του κράτους. Ε, ενώ οι πληρωμές πολλές φορές γίνονται μόνο με μετρητά. Κάποια άλλα ελληνικά συνέδρια αναφέρουν ότι ενδεχομένως κάποιες ομάδες συστηματικά μένουν εκτός της κάλυψης. Όλα αυτά είναι αδυναμίες οι οποίες εντοπίστηκαν. Έκτη πρόκληση, όπως λένε και οι συνάδελφοι του ΩΣΑ, υπάρχει ένα θέμα αποτελεσματικής παρακολούθησης της ένταξης ε, και της συνεπαγόμενης προσαρμογής των πολιτικών χρειάζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη πολιτικών οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες ανάγκες των μεταναστών. Όμως η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν απαιτεί από τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή να παρακολουθούν το αποτέλεσμα των πολιτικών. Το κατά πόσον δηλαδή η χρηματοδότηση βοηθάει τους μετανάστες να ενταχθούν στην πράξη ή όχι. Ένα τρίτο των κρατών μελών ανέφεραν ότι δεν διαθέτουν καθόλου δείκτες για να μετρήσουν το αποτέλεσμα των πολιτικών τους. Επίσης, διάφοροι φορείς, ε, εθνικοί φορείς μας ε, ανέφεραν πως ε, δεν υπάρχουν επαρκές πληροφορίες πολύ συχνά για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την ένταξη. Να πω εν παρενθέσει ότι αυτή η έλλειψη παρακολούθησης δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι της πολιτικής μας, αλλά γενικότερα της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η παρακολούθηση της απόδοσης των πολιτικών μας είναι πολύ σημαντικό θέμα οριζοντίως. Έβδομη πρόκληση, όχι λιγότερο σημαντική, εντοπίσαμε δυναμίες ό,τι αφορά την περιπλοκότητα των κανόνων χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, επιβάλλει στα κράτη-μέλη να έχουν συντονισμένους, μηχανισμούς συντονισμού για να αποφεύγουμε ε, επικαλύψεις, ε, αλλά δεν έχουν τέτοιους μηχανισμούς όλα τα κράτη-μέλη και μόνο τρία έχουν εκδώσει κατευθυντήρες γραμμές για συντονισμό. Χρειάζεται καλή, περισσότερη ηγετική δράση, ε, διότι τα ταμεία και η χρηματοδότηση γίνονται σε διάφορα επίπεδα και οι δαπάνε των ποσόνιων σε διάφορα επίπεδα, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό κλπ. Έχουμε πάνω από 400 διαφορετικέ αρχέ που εμπλέκονται στην διαχείριση των κοινοτικών πόρων για την ένταξη των ε, μεταναστών την περίοδο 2014-2020. Στην πολιτική συνοχή, μάλιστα, υπάρχουν άλλε 500 τέτοιε αρχέ και φορεί. Είναι δηλαδή πάρα πολύ πολύπλοκη αυτή η ιεραρχία. Χωρί επαρκή συντονισμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο υφίσταται ο κίνδυνο η περιπλοκότητα των ε, οικονομικών κανόνων να οδηγήσει σε μείωση της αποδοτικότητας του συστήματος. Αυτές είναι οι 7 προκλήσεις που εντοπίσαμε. Δεν εκδίδουμε συμπεράσματα, ούτε συστάσεις, διότι δεν πρόκειται για μια κανονική μας έκθεση ελέγχου, πρόκειται για ένα ενημερωτικό έγγραφο και λίγο πεπαλαιωμένο πια, όμως είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε αυτές τις δυσκολίες για να τις λάβουμε υπόψη μας στον πολιτικό μας διάλογο. Ευχαριστώ. Uh, ε, από όσο γνωρίζω υπάρχει μια κοινή παρουσίαση των δύο επομένων ομιλητών. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Έχετε ερωτήσεις για την κυρία Ιβάνοβα. Ε, παρέλειψα να πω ότι υπήρξε και ένα follow-up γιατί έκτοτε Είχαμε διάφορες εξελίξεις ε, με βάση το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής. Τότε έλειπαν 23 δράσεις, αλλά έκτοτε έχουν ολοκληρωθεί. Ως προς τη χρηματοδότηση, σας είπα ότι είμαι υπεύθυνη για θέματα συνοχής και υπάρχουν νέες προτάσεις ως προς την ένταξη. Τώρα το Ταμείο Ένταξης και Ασύλου θα ενταχθεί στα πλαίσια της συνοχής. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις για εσάς, αλλά θα μπορέσετε να παρέμβετε μετά από 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα για την εξαιρετική εργασία σε αυτό το έγγραφο ενημέρωσης. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η εργασία ήρθε την κατάλληλη στιγμή γιατί δημοσιεύθηκε η έκθεση όταν εγκρίθηκε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Επίσης, συμμεριζόμαστε τις απόψεις του ελεγκτικού συνεδρίου ως επιτοπλίστων. Θα ήθελα να τονίσω μερικές. Η διαδικασία ένταξης θα πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι η ένταξη έχει μεγάλη σημασία για την κοινωνική συνοχή τις κοινωνίες μας και γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν. Η κυρία Ιβάνοβα είπε ότι αυτό είναι ευθύνη κρατών μελών, αλλά η Επιτροπή πρότεινε βελτιώσει στα νομικά μέσα έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να αρχίζουν με την ένταξη σε προημότερα στάδια δηλαδή πρόσβαση των ετούντων άσυλο στην αγορά εργασίας έξι μήνες μετά την υποβολή της αίτησης και όχι εννέα όπως ισχύει μέχρι τώρα. Συμφωνούμε με το ελεγκτικό συνέδριο ότι χρειάζεται η χρηματοδότηση για να υπάρχει σωστή ένταξη και το επόμενο π δελτα πι θα ε, προωθήσει και το ΕΤΠΑ και τα διαρθρωτικά ταμεία για το ESF συν και τις βασικές προτάσεις. Ξέρετε ότι γίνεται αποκεντρωμένη διαχείριση και γι' αυτό θα πρέπει όλα τα ταμεία να εντάσσονται στην ε, αρχή της εταιρικότητας και να είμαστε σε επαφή με τις διαχειριστικές αρχές για να προβάλλουμε συγκεκριμένες εγγραφές κονδυλίων. Επίσης, θεωρούμε ότι χρειάζεται καλύτερος συντονισμός. Προτείναμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία και θα έχουμε μία κοινή παρουσίαση κατά τη συνάντηση του Ιουνίου. Θα συζητήσουμε με τις διάφορες διαχειριστικές αρχές για να έχουμε καλύτερη προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης. Επίσης, στην Κομισιόν έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση με τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιών για την καλύτερη χρήση των χρημάτων. Και τέλος, θα οργανώσουμε μία διάσκεψη κατά το τέλος του έτους, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ενημερώνουν εκείνους που εφαρμόζουν το πλαίσιο αυτό για να γίνει καλύτερη δυνατή χρήση των χρημάτων. Τέταρτον, συμφωνούμε ότι η πολιτική ε, ένταξη θα πρέπει να αφορά όχι μόνο τους πρόσφυγες αλλά και τους μετανάστες με οικογενειακές ανάγκες. Ε, επίσης, έχει μεγάλη σημασία η εποπτεία αυτού του καθεστώτος και δεν θα πω περισσότερα γιατί αυτό είναι το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όμως δεν συμφωνούμε με το ελεγκτικό συνέδριο ότι το πρόγραμμα εξαρτάται από τις εθνικές δεσμεύσεις γιατί το πρόγραμμα δράσης αφορά μέτρα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και όχι τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εστιάσουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτή η σύσταση όμως προαπαιτεί συγκεκριμένες δράσεις. Τέλος, η έκθεση βοήθησε ιδιαίτερα και συνεισέφερε στις σκέψεις μας για τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις, για την ένταξη και ελπίζω να έδειξα ότι υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο συμφωνίας με το ελεγκτικό συνέδριο και θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για αυτή τη χρήσιμη εργασία. Ο επόμενος ομιλητής... Κύριος Καρπέτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ε, ονομάζομαι Σκαρπέτα και με χαρά έρχομαι εδώ για να σας παρουσιάσω την ε, τελευταία δημοσίευση του κέντρου του ΩΣΑ για την απασχόληση, Διευθύνση Απασχόλησης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την ανακοίνωσή μας που θα βρείτε αντιγραφά της μάλιστα εδώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντα ότι η ανάγκη για παρακολούθηση που ανέφερε η κυρία Ιβάνοβα της ενσωμάτωση των μεταναστών στις χώρες αυτές εγγράφεται στο επίκεντρο της εκθεσή μας. Στην ε, προσεχή διαφάνεια λοιπόν, όπως είπα, κοινή προσπάθεια Ευρωπαϊκής Ένωση και όσα μακροπρόθεσμη και μακροχρόνια συνεργασία για να παρακολουθήσουμε και τις μεταναστευτικές ροές αλλά και την εξέλιξη που έχει η προσπάθεια για την ενσωμάτωση και ένταξη κοινωνία. Έχουμε λοιπόν μια πολύ συνολική εικόνα πιστεύω στην έκθεσή μας για την ένταξη στις κοινωνίες των χωρών των μεταναστών με χαρακτηριστικά που καταγράφουμε με εξέταση των επιδόσεων τους με βάση και τις, τα δικά τους χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα εξετάζουμε την ένταξη από διάφορε πτυχές, όχι μόνο δηλαδή στην αγορά εργασίας, αλλά ένταξη της πρώτης και δεύτερης γενιάς στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Η ιδιαίτερη αυτή λοιπόν έκδοση η νέα έκθεση του 2018. Έχει τρία επιπλέον κεφάλαια. Μια πτυχή που αφορά το φύλλο, διαφορά δηλαδή μεταξύ γυναικών και ανδρών, πάλι με βάση τα τα χαρακτηριστικά τους. Η ιδιαίτερη εστίαση δίνεται σε ένα άλλο κεφάλαιο στους νέους που προέρχονται από μεταναστευτικές οικογένειε μεταναστευτικών και μια άλλη πτυχή είναι αυτή που κάνει αναφορά σε πικόους τρίτων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τους δείκτες της Σαραγώσα. Θα ήθελα λοιπόν να κάποια στοιχεία. Βλέπετε εδώ στο γράφημα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της έχει έναν στους πέντε περίπου ε, που προέρχονται από γονείς είτε μετανάστευση είτε που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα. Βλέπετε τη διαφορά μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 30% σε ορισμένες χώρες όπως Ουγγαρία, Σλοβακική Δημοκρατία, Λουξεμβούργο ε, μέχρι 80% σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Κροατία και άλλες. Μεγάλη διαφορά λοιπόν και από το πού προέρχεται ο αλλογενής ε, πληθυσμός και πόσο είναι ο αλλογενής πληθυσμός. Ε, χαρακτηριστικά λοιπόν των αλλογενών ταξινόμηση σε δύο, στα δύο άκρα των δεξιοτήτων. Έχετε αριστερά τα, τις χαμηλές δεξιότητες σε σύγκριση ε, αναχώρα. Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία έχουν χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων πολύ μεγαλύτερο στους αλλογενείς από ότι στους ενδογενείς, ε, ηθαγενείς, ενώ στην άλλη πλευρά άλλες χώρες, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Σουηδία δείχνουν υψηλό ποσοστό δεξιοτήτων για τους αλλογενείς και ισοδύναμο ή αρκετά υψηλό σε σχέση και με αυτό των ηθαγενών. Έχουμε επίσης μια σημαντική αύξηση στην εισρωή νόμων μεταναστών με υψηλές δεξιότητες με αποτέλεσμα ο πληθυσμό των αλλογενών να τίνει να ε, παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων ε, συν το χρόνο. Αν και πάλι υπάρχουν αρκετές διαφορές με κατανομή ανάλογα με τις χώρε. Εδώ βλέπετε διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης, δηλαδή ποσοστό εκείνων που σε ηλικία ε, απασχόλησης παραγωγική έχουν μια θέση εργασίας ή αναζητούν συγγνώμη θέσει εργασία. Εδώ λοιπόν βλέπετε διαφορέ ανάλογα με τι χώρε, με το μπλε, έχετε τη διαφορά στην προσπάθεια στους, χαμηλέ ε, στις χαμηλές δεξιότητες. Στα δεξιά βλέπετε ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι που εργάζονται με χαμηλές δεξιότητες αλλογενείς σε σχέση με τους ηθαγενείς. Ενώ στο αριστερό κομμάτι βλέπετε ότι το χαμηλό επίπεδο της Αναζήτηση εργασίας στις χαμηλές δεξιότητες είναι υψηλότερο από ότι αυτό των ηθαγενών. Αριστερά βλέπετε τις χώρες που έχουν πολλούς πρόσφυγες και ε, δεύτερη γενιά μεταναστών, ενώ δεξιά βλέπετε κυρίως ε, νομιμοποιημένους μετανάστες. Και εδώ το επίπεδο απασχόλησης είναι χαμηλότερο όταν μιλούμε για ε, χαμηλές δεξιότητες σε σχέση με το ποσοστό των ηθαγενών. Η ένταξη βέβαια στις κοινωνίες ε, πολύ συχνά δεν αναγνωρίζει την, τις δεξιότητες. Έχουμε πολλούς, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια μετανάστες, των οποίων οι δεξιότητες δεν καταγράφονται σωστά ή δεν αναγνωρίζονται σωστά. Ε, και έτσι κάνουν δουλειές που απαιτούν πολύ χαμηλότερες δεξιότητες. Εδώ έχουμε τη διαφορά ε, στη μεταχείριση μεταξύ των φύλων, τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών. Το πιο ανοιχτό χρώμα είναι αυτό που αφορά τους ηθαγενείς, ενώ το ε, σκούρο χρώμα είναι αυτό που αφορά τους αλλογενείς και τις αλλογενείς μάλλον γυναίκες που έχουν γεννηθεί σε χώρες ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες και όταν μιλούμε για ένταξη η δυνατότητα μιας μητέρας να ε, λάβει μέρος στην αγορά εργασίας είναι και γεγονός που μπορεί να λαβει μερος στην αγορα εργασιας ειναι και γεγονό που μπορει να είναι καθοριστική σημασία για τα παιδιά της δεύτερης γενεάς και τη δυνατότητά τους και στο σχολείο να πάνε και αργότερα να σωματωθούν στην αγορά εργασίας. Η διαφορά λοιπόν στην αντιμετώπιση στα φύλλα έχει πολύ μεγάλη διαφορά στις αλλογενείς, ε, στους ε, πληθυσμούς αλλογενών γυναικών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του ΩΣΑ γενικότερα. Εδώ έχουμε εκείνους που έχουν γεννηθεί στην ε, χώρα, μεν προέρχονται όμως από αλλογενείς γονείς και η διαφορά είναι ε, στα ποσοστά απασχόλησης, αρνητική πάντα στις περισσότερες χώρες και πάντα με υψηλότερο το ποσοστό των χαμηλών δεξιοτήτων σχέση με τους ανθρώπους που έχουν υψηλές δεξιότητες. Ωστόσο, επειδή τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη φέρνουν καλά αποτελέσματα και έτσι καλύπτουν το χάσμα και το κενό ως προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση, παρόλα αυτά, ωστόσο, παραμένει ένα πρόβλημα γιατί τη στιγμή που μπαίνουν στην αγορά εργασία, οι δυνατότητε για εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν θα γεννή γεννημένος όμως από αλλογενείς γονείς ή μη. Και η επόμενη και τελευταία ουσιαστικά διαφάνεια, ουσιαστική διαφάνεια που έχω να σας δείξω έχει να κάνει με την αντίληψη σε σχέση με αλλογενείς ή ηθαγενείς, αν αισθάνονται δηλαδή ενσωματωμένοι ή μη στις χώρες υποδοχής. Και εδώ θέλω να ολοκληρώσω ότι με την παρουσίαση για να πω ότι είναι πολύ μικρές οι διαφορές, δηλαδή αλλογενείς ε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, 90% ε, αισθάνονται κατά 90% ότι έχουν θέση στην ε, χώρα υποδοχής τους μόνο 90%, δηλαδή μόνο 10% υπολείπεται από την αποδοχή που αισθάνονται οι ηθαγενείς. Και κλείνω με τελευταία διαφάνεια που σας δείχνει ότι οι υπηκοϊτροί των κρατών έχουν μια σειρά από εδώ πάλι για τις ε, διάφορες χώρες, ενσωμάτωση ως προς την απασχόληση, την ε, εκπαίδευση, κοινωνική ενσωμάτωση κτλ. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο της ε, μελέτης μας δίνει μια εικόνα των επιδόσεων των υπηκών τρίτων κρατών ως προς την ένταξή τους στις κοινωνίες των ευρωπαϊκών κρατών με σύγκριση των αποτελεσμάτων και αυτό το βλέπετε στα διαφορετικά χρώματα της διαφάνειας ανάλογα με τις χώρες του ΩΣΑ και σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν σχόλια, ερωτήσεις. Έχετε μείνει έξω όλοι, έτσι. Η κυρία Βεργιά. Ευχαριστώ πολύ και τους ναι και τους δε Είναι πολύ ενδιαφέρον να εργαζόμαστε σε συνολικά στοιχεία ανεξαρτήτως χώρας. Όμως όπως είδαμε υπάρχουν διακρίσεις ε, και αν μπορούσατε να μας δώσετε λίγο περισσότερα στοιχεία σε συνάρτηση με την χώρα προέλευσης ή την ήπειρο προέλευσης. Ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες διαφορές εκεί, αν δεν είμαι σωστά ενημερωμένη. Οι βασικέ χώρε προέλευσης σήμερα ε, των οποίων οι μετανάστε αυξάνεται με μεγαλύτερου ρυθμού είναι η Κίνα και η Ινδία. Προφανώ είναι οι πιο πολυπληθεί χώρε του κόσμου, οπότε είναι λογικό, αλλά έχετε εργαστεί με περισσότερη λεπτομέρεια στα στοιχεία έτσι ώστε να κάνετε διάκριση ανάλογα με τη χώρα προέλευσης σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις τι οποίε ε, τις οποίες υφίστανται οι μετανάστες. Okay, um, Κύριος Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ αν μου επιτρέπετε στα γερμανικά. Γιατί θα ήθελα να εκθέσω μια φιλοσοφική θεώρηση που έχει να κάνει και με την αγορά εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζει τα θέματα η κυβέρνηση της Αυστρίας. 30.000 δικαιούχοι ασύλου, νόμιμα δηλαδή μετανάστες, ε, που έχουν προσκληθεί, εκ των οποίων 1.800 προσκλήθηκαν σε μια αγορά, σε, μια σε ένα ανοιχτό φεστιβάλ ε, αγοράς εργασίας με πολύ καλή ανταπόκριση και θα ήθελα αυτό να το προτείνω όχι μόνο για τα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα ως ε, επίρρωση των ε, παρατηρήσεων της μελέτης σας, αλλά και ως φιλοσοφική θεώρηση για να πω ότι από το να έχουμε τους ανθρώπους αυτούς εξαρτώμενους από τα επιδόματα στο να συμβάλλουν στην κοινωνική ζωή και την οικονομική ζωή της χώρας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είπε άλλωστε ο καγκελάριος της Αυστρίας ότι δεν πρόκειται να φύγουν ούτε και θέλουμε να τους ξεφορτωθούμε. Θέλουμε να τους ενσωματώσουμε με τέτοια μοντέλα αλλά και με άλλα και έμαθα από εσάς τώρα και από πολλά σχέδια και πιλωτικά έργα που έχετε αναπτύξει, ότι πως υπάρχει αυτή η φιλοσοφία γενικευμένη και ότι είναι πολύ καλή. Έχει να κάνει λοιπόν με την προσφορά εργασίας και την αγορά εργασίας. Είναι πολύ καλό το ότι ενσωματώνεται και αυτή την διάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Σκαρπέτα. Καταρχήν, να Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσου είναι εδώ σήμερα. Η πρωινή συνεδρίαση ήταν πολύ κουραστική. Είμαστε όλοι εξαντλημένοι. Είναι χαρακτηριστική μέρα Επιτροπής ΛΥΜΠΕ με την αρχή τη Ρουμανική Προεδρίας. Όλοι μα είμαστε λίγο ζαλισμένοι. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν μειώνει την ποιότητα των, του έργου μας. η ένταξη είναι κρίσιμο ζήτημα και εμπίπτει, όπως και άλλα παρόμοια θέματα, στις δικές μας αρμοδιότητες, αλλά είναι και παγκόσμια και οριζόντια θέματα ταυτόχρονα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής για τη μελέτη του ΩΣΑ. Αν δεχτούμε ότι η ένταξη είναι ένα από τα πιο βασικά θέματα τα σχετικά με τη μετανάστευση. Και συμφωνήσουμε ότι θα χρειαστεί και στο μέλλον κάποιο είδους διαχείρισή της. Ε, είναι όμως ταυτόχρονα και ένα θέμα με πολιτικό φορτίο, πολιτικά φορτισμένο. Ε, η ερώτηση έχει λιγότερη σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά προς τον ΩΣΑ, που είναι ένα όργανο ε, γνωστό τό διάσημο, φημισμένο και σεβαστό όργανο. Όλοι σας σέβονται. Αισθάνεστε ποτέ, αισθανθήκατε καθόλου ότι ε, ασχολούμενοι με θέματα ένταξης θα έπρεπε να δείτε καλύτερα τι πραγματικότητε της μετανάστευση και τη ένταξη. Χωρίς να το λέω με κακό τρόπο. Στο τέλος όμως λέτε... Ε, όταν μιλάτε για διακρίσεις, ε, ε δεν λέτε διακρίσεις, λέτε αντιληπτές ως διακρίσεις. Ε, γιατί δεν το λέτε ξεκάθαρα. Ε, πρόκειται για ρατσισμό, πρόκειται για μίσος. Είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των συγκρούσεων που βλέπουμε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή δεν αναθεωρεί την οδηγία για την μπλε κάρτα ε, και ε, δεν είναι ε, πολύ περίπλοκα τα επιχειρήματα αυτών που αρνούνται. Είναι πολύ απλά, δεν θέλουν οι Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τέτοιες αρμοδιότητες, γιατί φοβούνται. Εσείς τον όσα αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάτε. Μιλάμε για διαφορετικές φυλές, διαφορετικές εθνότητες, δεν πρόκειται για οικονομικό μόνο θέμα. Και Οπότε εσείς κοιτάτε δείκτες όπως ε, προβλήματα στέγαση, ανεργία κλπ. Αλλά είναι λίγο σχιζοφρενικό, διότι ε, έχουμε τεράστιους πληθυσμούς που καταλαβαίνουν ποια είναι τα προβλήματα. Καταλαβαίνουν ποιο είναι το πρόβλημα ε, αυτό είναι το πρόβλημα. Των διακρίσεων του μίσου του φόβου. Οπότε η ερώτησή μου είναι πώς το βλέπετε εσείς αυτό τον παράγοντα τον οποίο δεν καλύπτεται με τους δείκτες. Όσα είναι σεβαστός από όλους ο οργανισμός ε, και ασχολείται με δημογραφικά και με οικονομικά στοιχεία, με την οικονομική διάσταση, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τι βρίσκεται μάλλον στο επίκεντρο του προβλήματος της ένταξης. Γιατί οι τοπικές κυβερνήσεις κάνουν αυτά που κάνουν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύεται τόσο πολύ, γιατί, γιατί τα διαχειριζόμαστε με τόσο κακό τρόπο αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. το σκεφτόσαστε καθόλου όλο αυτό. Εσείς λέτε perceived discrimination. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει διάκριση, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για αντιληπτή ως διάκριση. Αυτή την έκφραση χρησιμοποιούν κάποιοι οποίοι δεν θέλουν να μιλούν για διακρίσεις. ενδεχομένως αποφεύγετε να μιλήσετε για αυτό το θέμα με καθαρούς όρους για να μην φοβήσετε. Αλλά ο λόγος για την ένταξη είναι επειδή οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Οπότε αναρωτιέμαι μήπως κάποιοι οργανισμοί, μεγάλοι οργανισμοί και φορείς βλέπουν το θέμα μόνο από οικονομικής και δημογραφικής πλευράς, αλλά υπάρχει απόσταση από την πραγματικότητα και ίσως αν κλείναμε αυτή την απόσταση, αυτό το κενό, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να, περάσουμε, να, να παρακάμψουμε, να υπερβούμε και τα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω των οτροπιών μας. όλα αυτά τα σκέφτηκα βλέποντα αυτή την έκφραση, το perceived discrimination. Δεν ξέρω, εσεί το εντοπίσατε αυτή, την, αυτή την, τη λέξη. Όχι μόνο την εντόπισα, ε, ε, αλλά είναι επίτηδε εκεί. Θα σα εξηγήσω. Καταρχήν, χωρίς προέλευση. Αν δείτε αυτή τη δημοσίευση, αλλά και τη δημοσίευση για, την, για το πανόραμα της διεθνής μετανάστευσης, ασφαλώς και εξετάζουμε τις χώρες προέλευσης. Ε, για κάθε μία από τις χώρες υποδοχής έχουμε ροές από διάφορες χώρες προέλευσης. Ο κύριος Μπέκερ απευθύνθηκε πιο πολύ στην Κομισιόν, έχει δίκιο, αλλά να πω το εξής. Ο, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, των εργοδοτών της κοινωνίας των πολιτών ε, στην ένταξη ιδιαίτερα στην ένταξη των μεταναστών, ε, προσφύγων. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα εμπόδια τα οποία θεωρούν ότι υπάρχουν οι εργοδότες και γι' αυτό το λόγο δεν τους προσφέρουν απασχόληση. Στη Γερμανία, ας πούμε, οι εργοδότες θέλουν να αποτέλεσουν τμήμα της λύσης, αλλά θέλουν πολύ θέτουν πολύ συγκεκριμένους όρους στην κυβέρνηση. Τώρα, για τη δική σας ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Ε, το, η διαφορά ανάμεσα στα στατιστικά, τα νούμερα αφενός και την αντίληψη που έχουν ε, ε οι άνθρωποι. Ε, ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποίησαμε αυτό τον όρο είναι διότι ρωτούσαμε τους ανθρώπους αισθάνεστε να γίνετε διάκριση εναντίον σα όταν προσπαθείτε να μπείτε στην αγορά εργασία. Αυτό είναι ένα γιατί το αισθάνονται και άλλο η πραγματική διάκριση που μπορεί να γίνει ε, εκ μέρου των εργοδοτών. Πάντω είναι πολύ σωστό το επιχείρημά σα. διότι αυτή τη στιγμή ε, ετοιμάζουμε μια πιλωτική μελέτη για να εντοπίσουμε τα στατιστικά εργαλεία που χρειάζονται για να εντοπίσουμε την πραγματική, τις πραγματικές διακρίσεις. Για παράδειγμα, τυφλή πρόσληψη, όπου στέλνουμε χωρί ο εργοδότη να το ξέρει άτομα με τα ίδια προσόντα αλλά από διαφορετικέ εθνότητε για να δούμε αν ο εργοδότη θα κάνει διάκριση ή όχι. Ε, έχω μια ιστορία, ένα παρελθόν στην ε, ε, Επιτροπή ε, Κοινωνικών Θεμάτων. Στην πράξη με ελάχιστε εξαιρέσει, καμία χώρα δεν έχει εφαρμόσει πραγματικά την νομοθεσία για την ε, αποφύγη των διακρίσεων στην αγορά εργασία. Δεν έχουμε καν δεδομένα. Οπότε αυτό που είπατε εσεί για τυφλή δοκιμή ε, έχει γίνει ήδη και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά ανησυχητικά. Είναι ε, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε, στο 50% των περιπτώσεων γίνονται αρνητικές διακρίσεις με βάση την προέλευση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει εργασία, εργασιακή, εργατική νομοθεσία για αυτά τα θέματα, οπότε δεν πρόκειται να βρείτε δεδομένα, δεν πρόκειται να βρείτε στοιχεία αριθμητικά. Όταν μιλάμε για διακρίσεις, δεν εφαρμόζεται η οδηγία ισότητας, για παράδειγμα, Ο βασικός δείκτης ε, είναι η διαφορετικότητα. Διαφορά στη γλώσσα, διαφορετικά στη διαφορά στη χώρα προέλευση κλπ. Οπότε πολύ καλά κάνετε τη δουλειά σας, αλλά όσο προχωράμε, τόσο πολύ θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα και δεν έχουμε τα εργαλεία. Και βέβαια, οι κακόβουλοι λαϊκιστές κλπ. Έχουν πάει πολύ πιο μακριά από εμά και καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα τη φύση του προβλήματος και γι' αυτό το λόγο κάνουν ζημιά. Γι' αυτό το λόγο είναι και επίγον να κάνουμε και εμείς τη δική μας δουλειά. Χρησιμοποιείτε άλλου δείκτε, στου οποίου είστε πάρα πολύ καλοί, δείκτε ανεργία κλπ. Αλλά λάβετε υπόψη και αυτό που λέω, μη με παρεξηγήσετε. Ωραία να ρωτάτε τον άλλο αν πιστεύει ότι υφίσταται διακρίση, αλλά δεν αρκεί. Πολύ σωστά αυτά που λέτε, λέει ο κ. Σκαρπέτα. Σίγουρα ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα, τα στοιχεία, για να τροφοδοτήσουμε μια δημόσια, ένα δημόσιο διάλογο. Τα νούμερα είναι πολύ ε, σαφή. Ίσως δεν έχουμε στοιχεία για τα πάντα, αλλά αν συνδυάσουμε αυτά που έχουμε, θα δούμε διαφορά στα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την απασχόληση, τον τύπο δουλειά, τους μισθούς κλπ. Εκεί μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Οπότε εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα δεδομένα μας μπορούν να μας πούν για παράδειγμα ποιες χώρες τα πάνε καλύτερα, ποιες πολιτικές είναι οι καλύτερες, ποιες κοινότητες τα πάνε καλύτερα και κάνουν περισσότερες προσπάθειες ένταξης. Το σημαντικό όμως είναι το netcom, δηλαδή το δίκτυο των ανθρώπων, αξιωματούχων, ανώτερων αξιωματούχων, που συζητούν μεταξύ τους για το πώς μπορούν να αλληλοενημερώνονται για τις πολιτικές τους και το πώς μπορούν να αντιδρούν στα σαν αναφέρονται στα μέσα ε, μαζικής ενημέρωσης λοιπά στα, στα διάφορα ψεύδη ή τα λαϊκιστικά επιχειρήματα που αναφέρονται. Εμείς έχουμε πολλά στοιχεία, πολύ σαφή και πολύ ρητά και πολύ κατηγορηματικά, αλλά πολλές φορές η συζήτηση πηγαίνει προς άλλη κατεύθυνση στις χώρες μας. Οπότε ε, σίγουρα χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα, αλλά δεν είναι αρκετό βέβαια. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα το πώς αισθάνονται και πώς σκέφτονται οι πολίτες μας. Ίσως μέσω του Ευρωβαρομέτρου θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να δούμε τι είναι αυτό που ανησυχεί πιο πολύ τους πολίτες μας. Είναι πολύ καλά τα νούμερα του ΩΣΑ. Και συγχαρητήρια στην Κομισιόν που πιέζει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, την οδηγία για την ισότητα, παρόλο που δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου. Μπορώ να πω και ονόματα κρατών που δεν ε, εφαρμόζουν την νομοθεσία. Έχουμε αρκετά λεπτομερή στοιχεία Είναι σαφές ότι κάποιες χώρες είναι καλύτερες από κάποιες άλλες, αλλά η κατάσταση είναι πολύ απλή μάλλον είναι πολύ, πολύ φτωχή σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για την ένταξη. Ο κ. Νάκη δεν είναι εδώ ακόμα. Ε, δεν προσπαθούσα να καθυστερήσω. <laughs> Δεν έπαιζα καθυστερήσεις. Ήταν σοβαρό αυτό που έλεγα. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. για το Ελεκτικό Συνέδριο. Χαίρομαι που έχουν εκδοθεί όλες αυτές οι, οι εκθέσεις για το άσυλο, τη μετανάστευση κλπ. Ε, εστιασμένες. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ το Ελεκτικό Συνέδριο για όλα αυτά τα ενημερωτικά έγγραφα και ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους από την Κομισιόν και από τον ΟΣΑ, τον κύριο Σκαρπέτα, για, για, για παράδειγμα. Ευχαριστούμε κύριε Μπέκερ, Μαρή Κριστίν κλπ.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 Sorry, I know this is testing everyone's patience today, but our... Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι δοκιμάζω την υπόμονη όλων σας. Σε 5-10 λεπτά ξεκινάει το επόμενο θέμα, όταν έρθει ο κύριος Νάγκη του. Ζητήσαμε βέβαια να έρθει πιο νωρί για να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε όσο το δυνατόν πιο νωρί. Είναι καθοδόν. Και εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και κυρίως τους βουλευτές και το προσωπικό μας που είναι εδώ και περιμένει.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 Uh, sorry, colleagues. Let's get started. Ας ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι και το τελευταίο μας θέμα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Έχουμε ένα σχέδιο σύστασης στη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης για το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη εξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Ιώζεφ Νάγκη, Ολοκληρώνει την διαπραγμάτευση επί τετραετία του πρωτοκόλλου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, προετοιμάζει προσκύρωση το πρωτόκολλο. Με χαρά δίνω το λόγο τώρα στον εισηγητή κύριο Νάγκη. Και τον ευχαριστώ που ήρθε και λίγο νωρίτερα. Μπορείτε να λάβετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο εισηγητής θα ήθελα να συστήσω την, να σχολιάσω καλύτερα την πρόταση για σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου στο πρωτόκολλο για την τροποποίηση της σύμβασης του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης για την ε, προστασία των ατομών σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, ETS αριθμός 108. Η τροποποίηση λοιπόν του πρωτοκόλλου ξεκίνησε παράλληλα με τη μεταρρύθμιση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη δέσμη μέτρων δηλαδή συμπληρωματικό εργαλείο, αντικατοπτρίζει τη σχετική νομοθεσία, το GDPR και την οδηγία για τα δεδομένα στην αστυνομία. Η σύμβαση αυτή λοιπόν 108 έχει κρίσιμο ρόλο για την στήριξη του προτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συχνά είναι μάλιστα και πηγή έμπνευσης για χώρες που αποφασίζουν να ε, αναθεωρήσουν ή να εξυγχρονίσουν με διεθνείς προδιαγραφές την νομοθεσία τους για τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι λοιπόν διευκολύνεται η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με βάση κοινέ ε, ασφαλιστικές δικλείδες, διευκολύνει την ροή δεδομένων, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση αλλά και κρατών εκτό Ευρωπαϊκής Ένωση που είναι συμβαλόμενα μέρη στη σύμβαση εισάγει τη δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλους διεθνεί οργανισμούς να καταστούν συμβαλόμενα μέρη στη σύμβαση και σας ευχαριστώ. 28 Ιανουαρίου κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ, Ιώζεφ. Η Επιτροπή. Ο κύριος ε, Φρανς που περιμένει τόσο υπομονετικά. Φρανς. Σκιώδης. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ έχουμε ακόμα ένα παράδειγμα του πώς η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έχει διατυπωθεί σωστά έχει διεθνή αντανάκλαση. Η Σύμβαση λοιπόν 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, ήδη από το 1980 υφίσταται και έχει αποτελέσει μάλιστα την πρώτη οδηγία ή την έμπνευση για την πρώτη οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων το 1995. Τώρα όμω η κατάσταση αυτή αντιστράφηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει με τον Φίλιπ Άλμπρεχτ και την προσήλωσή του, αλλά και των λοιπόν συναδέλφων των άλλων πολιτικών ομάδων, με την ε, προσπάθεια για την υιοθέτηση ενό κανονισμού για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων που ετέθησε ισχύ πέρυσι. Αυτή η ανανεωμένη μορφή λοιπόν τη ε, Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη έχει σε μεγάλο βαθμό ακολουθήσει το μοντέλο αυτού του κανονισμού GPRS, η μεγάλη συμμετοχή ε, και κρατών μάλιστα εκτός της Ευρώπης ε, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης δείχνει πόσο μεγάλο αντίκτυπο μπορεί να έχει το έργο μας ε, και πέραν της Ευρώπης σε ολόκληρο τον κόσμο. Το καλωσορίζουμε. Εμείς λοιπόν οι πράσινοι χαιρετίζουμε την ε, ενσωμάτωση με τη μορφή αυτού του πρωτοκόλου της αναθεώρησης της Σύμβασης 108 και ελπίζουμε και οι Ηνωμένε Πολιτείε να ενσωματωθούν στο, στη σύμβαση αυτή γιατί υπάρχουν ε, μεταξύ άλλων πολιτείες όπως η Καλιφόρνια που για πρώτη φορά βλέπουμε να υιοθετεί ένα διεξοδικό νομοθέτημα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε κάτι να προσθέσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουμε τις αξίες μας όπως ελέγχθη η σύμβαση ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων αλλά έχουμε 53 συμβαλόμενα μέρη ε, δηλαδή πολύ πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κινείται αυτό το μέσο και το σύμφωνο στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, έχουμε συμμετέχοντες και παρατηρητές στην ε, Ασία. Ελπίζουμε να έχουμε και το πρώτο συμβαλόμενο μέρος από την Ασία και θεωρώ ότι αυτό το μέσον μπορεί να προωθήσει τα δικά μας πρότυπα προστασίας δεδομένων ανά τον κόσμο. Τον Ιανουάριο του 2017 στην ανακοίνωσή μας μιλήσαμε για μια στρατηγική προστασίας και ροής δεδομένων. Και υπήρξε και ένα πλαίσιο για έναν κανονισμό περί ιδιωτικότητας στις ΗΠΑ και εμείς ζητήσαμε από τις ΗΠΑ να συμπλεύσουν και να προσχωρήσουν με τη Σύμβαση 108. Η ΕΠΑ αυτή τη στιγμή θέλει να προωθήσει το APEC, ένα εναλλακτικό μοντέλο σε σχέση με τους κανόνες ιδιωτικότητας ε, δυστυχώς με πολύ χαμηλότερες προδιαγραφές, αλλά νομίζω ότι το σύμφωνο 108 είναι ένα μέσον με το οποίο μπορούμε να ανταγωνιστούμε, να συναγωνιστούμε. Έχει κυρωθεί, αλλά αυτό είναι το πρώτο βήμα και για να τεθεί σε ισχύ χρειάζεται 38 συμβαλόμενα μέρη τα οποία θα πρέπει να κυρώσουν τη συμφωνία. Έχει αρχίσει η κυρωτική διαδικασία. Έχουμε 10 κράτη-μέλη που δεν έχουν καν υπογράψει τη σύμβαση. Προσπαθούμε να το προωθήσουμε με τα κράτη-μέλη. Και ίσως και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν δίνοντας το καλό παράδειγμα. Τη στιγμή που υπάρχουν συγκρίσιμοι κανόνες, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπογράψουν αυτό το μέσον και όταν δοθεί το πράσινο φως ε, κύρωσης, τότε θα κυρωθεί πολύ γρήγορα. Διαφορετικά θα περιμένουμε πολλά χρόνια μέχρι να τεθεί σε ίσχυ και θα ήταν πολύ κρίμα γιατί ήταν πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Τζόζεφ, θέλεις να επανέλθεις. Όχι. Στις 20 Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι τροπολογίες. Είναι η προθεσμία. Γεια σας. Καλό βράδυ. Αρχίσαμε, ε, τελειώσαμε λίγο νωρίτερα. Θα σας δω αύριο το πρωί. Γεια σας.